Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται. Τα συνοπτικά πρακτικά και τα κείμενα που εγκρίθηκαν στην χθεσινή συνεδρίαση έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις? Δεν φαίνεται να υπάρχουν, οπότε τα συνοπτικά πρακτικά εγκρίνονται. Τώρα η ημερήσια διάταξη προβλέπει δηλώσεις